Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Καλώ ήρθατε σε αυτή τη δεύτερη μέρα συνεδρία της Υποεπιτροπή ΕΝΤΕ. Σήμερα θα συζητήσουμε για τις συνέπειες του Brexit και την κατάσταση μετά το Brexit και τις πολιτικές που αφορούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Καλώς ήρθατε και πάλι. Να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε πολύ πεισμένοι χρονικά σήμερα το πρωί, γιατί μετά τα δύο πρώτα σημεία της ημερήσιας διάταξης που αφορούν το Brexit θα πρέπει να σπεύσουμε, ελπίζω να μείνουμε όλοι. Στο άλλο κτίριο, στο κτίριο Αλτιέρα Σπινέλη, στην αίθουσα 3Ε2, εκεί Έχουμε το στρατηγικό διάλογο με την ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μογκερίνη. Σε κοινή συνεδρίαση με τις επιτροπές ΑΦΕΤ και ΤΡΟΑ. Θα γίνει μάλιστα και κλεισμένο των θυρών. Και θέμα θα είναι τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα. Οπότε μετά το πρώτο μισό της συνεδρίασης θα μεταβούμε στην 3ε2 για το στρατηγικό διάλογο και θα επιστρέψουμε εδώ στις 11 με 12.30 για τη συνέχεια της ημερήσιας διάταξής μας. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι λοιπόν και στην ε, άλλη συνεδρίαση και μετά πάλι εδώ πίσω. Είναι κάπως περίπλοκο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Θα ακούσουμε τώρα την παρουσίαση μιας μελέτης ε, που την αναθέσαμε στην Επιτροπή στο Τμήμα Πολιτικής ε, στο Τμήμα Πολιτικών από τους συντονιστές ε, και το διευρυμένο Προεδρείο της ΕΝΤΕ με θέμα ε, πώς θα διαμορφωθεί κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας μετά το Brexit και τη μέλη γενέστε. Με ιδιαίτερη χαρά θα δώσω το λόγο στον ε, συντάκτη αυτής της μελέτης, στον εισηγητή, τον κύριο Φεντερίκο Σαντοπίντο, που εκπροσωπεί το GRIP. μια οργάνωση που συμμετείχε και χθε στη συνεδρίαση. Κύριε Σαντοπίντο, έχετε το λόγο. Μην επεκταθείτε πολύ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άμα επιτρέπετε, θα μιλήσω γαλλικά. Κυρίες και κύριοι, εξότιμοι ευρωβουλευτέ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης που κάναμε στο GRIP για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα και τον Brexit. Πριν περάσω στο κυρίω θέμα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία ως προ το υπόβαθρο. Ονομάζομαι Φεντερίκο Αντοπίντο, είμαι ερευνητή στο GRIP. Ε, Πρόκειται για ένα γαλλόφωνο ερευνητικό Ινστιτούτο μέτρα τη Βρυξέλλε και εγώ ασχολούμαι με θέματα άμυνα και εξωτερική πολιτική. Ενώ το κρύπτο το Ινστιτούτο μου ειδικεύεται κυρίω σε θέματα με ε, έλεγχο όπλων, ε, παρουσία τη ε, ένοπλη σύραξη και το καθεξή. Το Ίδρυμα για τη Στρατηγική Έρευνα, που είναι ένα γαλλικό ίδρυμα, έχει συνάψει σύμβαση πλαίσιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να εκπονεί συγκεκριμένε μελέτε για θέματα που άπτονται τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλεια και Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μα ζήτησε να εκπονήσουμε μία ανάλυση για τον Brexit και την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα με τίτλο CSDP μετά τον Brexit, τη μέλη γενέστε. Στα πλαίσια τη μελέτη αυτή, ε, αναλύσαμε σε μια πρώτη φάση τη βρετανική θέση και κυρίως ε, τις προτάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία. Και στη συνέχεια μας ζητήθηκε να εξετάσουμε τον αντίκτυπο του Brexit και τη νέα σχέση που προτείνουν οι Βρετανοί στα πλαίσια των μελλοντικών σχέσεων ε, στην κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας. Δεν πρόκειται να σας δώσω πολλά νούμερα για τη συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ασφάλεια και την άμυνα. Ε, γιατί αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, ήδη πρόσφατα δημοσιεύτηκαν από μία μελέτη της Κλίνκενταλ. Οπότε δεν χρειάζεται να καταιγιστείτε από στοιχεία. Και σε ό,τι αφορά την πολιτική ασφάλεια και άμυνας, ε, πριν ε, οι Βρετανοί αποφασίσουν την αποχώρησή τους, ήδη είχαμε φτάσει σε νεκρό σημείο στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οπότε έπρεπε να απεμπλακεί η κατάσταση και να αλλάξει κάτι, γιατί ε, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε έτσι. Οπότε μας δημιουργεί κάποια σύγχυση ότι παρουσιάζεται ως τραγωδία ή ως δράμα το Brexit. Κάτι έπρεπε να γίνει πριν κάτι αλλάξει βέβαια η σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο για, το, για την ασφαλεία και άμυνα. Βέβαια το Brexit ε, έχει προκαλέσει αναστάτωση στο τοπίο και θα πρέπει να γίνει μια αναδιάταξη και θα ήταν όμως παράλογο να προσπαθήσουμε απεγνωσμένα να αποκαταστήσουμε τις ισορροπίες του παρελθόντος ή να τις αναπαράγουμε. Γιατί αυτές οι ισορροπίες ήταν που μπλόκαρα για πολύ καιρό την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας που είχε μείνει σε σημείο νεκρό για πολλά χρόνια. Οπότε δεν θα πρέπει να θεωρούμε τραγωδία το Brexit. Οι αναλυτές και οι ερευνητέ όπως εγώ, μερικές φορές ε, δεν θέλουμε να φύγουμε από την άνεσή μας, από τη βολή μας και φοβόμαστε τις ρηξικέλευτες πολιτικές αλλαγές. Ιδιαίτερα όταν είναι απροσδόκητες, όταν ε, δεν προβλέπουμε κάτι, το, τίνουμε να το αντιμετωπίζουμε ως καταστροφή όταν συμβαίνει. Γιατί συχνά καταστροφολογούμε. Και μάλιστα αυτό σε αυτό ειδικεύονται οι οικονομολόγοι. Πόσε φορέ δεν μα ανήγγειλαν τη συντέλεια του κόσμου, ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τι οικονομικέ συνέπειε του Brexit. Αλλά και οι αναλυτέ που ασχολούνται με θέματα ασφάλεια και άμυνα είναι επίση ε, καταστροφολόγοι. Έχουν μια ροπή προ την καταστροφολογία. Ε, βέβαια, η μελέτη θέλει να κρύψει τα προβλήματα που δημιουργεί το Brexit ε, για την Ευρώπη γενικώ και την κοινή πολιτική άμυνας από ασφάλεια και άμυνα, γιατί είναι τεράστιο το διακύβευμα και πολύ σοβαρέ συνέπειε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική συνεργασία και την ανάπτυξη των μελλοντικών οπλικών συστημάτων. Οπότε οι διαπραγματεύσει του Brexit ε, είναι όντω επικίνδυνο ζήτημα. Αλλά ο τολμονικά. Και σίγουρα πολλά πράγματα έπρεπε να αλλάξουν στα πλαίσια της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. Οπότε παρά τους ορατούς και πραγματικούς κινδύνους ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Brexit θα είναι και ευκαιρία. Θα δημιουργήσει και ε, προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ευκαιρία γιατί το σχέδιο Ευρωπαϊκής Άμυνα που θα πρέπει να περάσει από μια φάση συνεργασία σε μια ουσιαστική φάση ολοκλήρωσης θα πάρει μια νέα πνοή και αυτό φαίνεται ότι έχει γίνει. Και άλλη ευκαιρία είναι γιατί μακροπρόθεσμα και όλος παραδόξος το Brexit μου λένε να επιβραδύνω κάπως γιατί φαίνεται ότι μιλάω πολύ γρήγορα Όλο παραδόξω, το Brexit μπορεί να βελτιώσει και όλα στη συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μέχρι στιγμή ήταν πολύ μέτρια. Οπότε δύσκολα να επιδεινωθεί η κατάσταση. Και ίσως απέναντι στο Brexit το Ηνωμένο Βασίλειο ενδιαφερθεί για πιο ενεργή συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα. Γιατί από τότε που αποφάσισαν τον Brexit, οι Βρετανοί δεν ήταν ποτέ τόσο επικοδομητική και δεν έδειξαν τέτοιο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή άμυνα. Ίσως ε, τώρα κατάλαβα την αξία τους με τον κίνδυνο να τη χάσουν. Οπότε πέρασαν από το, από το σκεπτικισμό σε ε, κάποιον που ζητά περισσότερη άμυνα, που όμως έχει χάσει το δικαίωμα αρνησή κυρίας τους, κάτι που ευνοεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για να αντιληφθούμε τις μελλοντικές σχέσεις που θα έχουν οι Βρετανοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην άμυνα, δεν αρκεί να ε, εξετάσουμε μόνο τις επίσημες προτάσεις. Θα πρέπει να δούμε γιατί ξαφνικά άρχισαν να εγκομιάζουν τόσο την κοινή πολιτική ασφάλεια και, ασφάλειας και άμυνας. Ίσως το ενδιαφέρον τους εξηγείται από το φόβο της περιθωριοποίησης μετά το διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα σε περίπτωση που εγκαταλείψουν και την Τελωνιακή Ένωση και την Ενία Αγορά. Οπότε βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παράδοξο. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Άμυνα θα είναι ο συνδετικό ιστό ουσιαστικά που θα συνδέσει τι Βαρδανικέ νήσου με την ε, υπηρετική Ευρώπη. Κάτι που ήταν το βασικό πρόβλημα ε, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η στάση του, Ευρωπαϊ... του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά δεν είναι το μόνο παράδοξο. Το νέο, η νέα ευρωπαϊκή άποψη ε, και το βλέμμα τους προς την ευρωπαϊκή άμυνα εξηγείται και από τι γεωπολιτικέ ανακατατάξει. Ε, που έφεραν ε, οι εκλογές ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και η ανάδειξη του Πρόεδρου Τραμπ και η αναστάτωση της σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί αυτές οι σχέσεις στηρίζονται σε μια αδιάστη εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία του εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών και στο ΝΑΤΟ και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η γεωπολιτική πολιτική επίσης ε, του Ερντογκάν, του Τούρκου Προέδρου, δημιούργησε κάποια αστάθεια και η γαλλική πρόταση για την εξασφάλιση μιας στρατηγικής αυτονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Και σίγουρα αν η αξιοπιστία των είπα είναι αυτόματη και αν το ΝΑΤΟ μπορεί να παραλύσει λόγω της Τουρκίας, ε, ε, φαίνεται ότι οι Βρετανοί χρειάζονται ε, όχι μόνο ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Σε ό,τι αφορά την Ιρανική Συμφωνία ή τι κλιματικέ αλλαγέ, κατάλαβαν ε, με την επαναχώρηση του Τραμπ. Επίση, ε, άλλο παράδοξο, γιατί το Brexit είναι πραγματικά ένα μεγάλο παράδοξο, φαίνεται ότι περισσότερο από ποτέ το Λονδίνο χρειάζεται την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Από το 1998 που πρωτοτέθηκα τα θεμέλια τη. Ποια είναι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, απλούστατη. Οι αρμόδιε αρχέ τη χώρα θέλουν ε, ενεργό εμπλοκή στο μέτρο του δυνατού στην πολιτική ασφάλεια και άμυνα και στη βιομηχανική πτυχή και στην επιχειρησιακή πτυχή τη ε, πολιτική. Αν εξαρτάταν από του Βρετανού μόνο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα έμενε ακέραιο μέλο, πλήρε μέλο και τη ΠΕΣΚ και τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Αυτό ίσω λόγω σύνεση ε, και επιφυλακτικότητα δεν αναφέρθηκε, αλλά έχει επισημανθεί και στη, στη, διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πάντως η ιδέα ότι το Brexit θα πρέπει να έχει το λιγότερο δυνατό αντίκτυπο, έως και μηδενικό αντίκτυπο στη συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, δεν ε, εμφανίζεται αυτή η ιδέα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε πολλές ομάδες σκέψης και προβληματισμού και στην αμυντική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή είναι η γνώμη που, έχουν και, που είχαν και οι οργανωτές της ε, ε, διάσκεψης του Μονάχου ε, του, με τίτλο «Να κρατήσουμε την Ευρώπη ασφαλή και μετά το Brexit». η πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή και τον παρακαλεί να μιλάει λίγο πιο αργά. Μετά από μια διακήρυξη που, που έχουν υπογράψει ο Ντασό, Κίσιγκερ και άλλοι επιφανείς του κλάδου. Το ενδεχόμενο λοιπόν να παραμείνω στο δυνατόν πιο κοντά στην κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα τη Ένωση οι Βρετανοί δεν φαίνεται κάποια χιλιόμετρα πιο πέρα στι εγκαταστάσει να, να έχει ιδιαίτερη απήχηση και θα πρέπει να καταλάβουμε για το τι μιλάμε. Και υπάρχουν κάποιε παρανοήσει. Συμφωνούν όλοι ότι η ανάγκη με το Λονδίνο να ε, διατηρηθεί όσο το δυνατόν πιο στενή συνεργασία σε θέματα άμυνα και ασφάλεια είναι προτεραιότητα. Όλοι θέλουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία με τους Βρετανούς. Εκεί όμως που υπάρχει μια βαθιά παρανόηση είναι η πρόσβαση που θα πρέπει να έχει ε, στις ε, σωρές λήψη αποφάσεων τη ΚΕΠΑ και τη ΚΕΠΑ η Βρετανία. Και εκεί είναι η όλη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφυλακτική και διστακτική απέναντι στις περισσότερες αναλύσεις. Φυσικά είναι ανοιχτή ε, στην ιδέα ε, και θέλει να υπάρχουν μηχανισμοί διαβούλευσης. Το λέει και η έκθεση μετάβασης, αλλά ε, έχει περιορίσει τις φιλοδοξίες των, και τις προστοκίες των Βρετανών ως προς το ότι θα χαίρουν ένα ειδικό καθεστώς παρατηρητή στις, στα βασικά όργανα δηλαδή Συμβούλιο και κόψ της ε, κοινή πολιτικής και είναι επιφυλακτική η Κομισιόν στην ιδέα του Λονδίνου να ενταχθεί στις δομές που θα αναλάβουν τη διαχείριση νέων πρωτοβουλειών ε, που έχουν μεγάλη σημασία στο βιομηχανικό τομέα, όπως το European Defense and Industrial Development Program, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ή την ε, συντονισμένη ή μάλλον τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Κατά περίπτωση και κατά σχέδιο θα πρέπει να γίνεται αυτό και όπως ε, πρεσβεύει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να υπάρχει κοινή διαχείριση των εν λόγω προγραμμάτων σε στρατηγικό και πολιτικό επίπεδο. Αυτή είναι η θέση της Κομισιόν αλλά και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου φυσικά. Και έχει παγώσει ουσιαστικά κυριολεκτικά τους Βρετανούς και έχει αφήσει επίσης ε, προβληματισμένους και τους ε, γενικότερους σχολιαστές του θέματος. Δύο διαφορετικές σχολές ε, έχουμε για το πώς πρέπει να σχετιστεί στο μέλλον η Βρετανία στην κοινή πολιτική ασφάλεια και άμεση και βιομηχανική τεχνολογική πολιτική. Η πρώτη σχολή υποστηρίζει την αρχή ότι το Λονδίνο θα πρέπει να είναι το δυνατόν πιο στενά συνδεδεμένο στις διαδικασίες της ΚΕΠΑ και της ΚΕΠΑ. λόμπι, ε, βιομηχανική πολιτική, think tank κτλ. Δεύτερη θέση, δεύτερη σχολή, επιφυλακτική, διστακτική να παραμείνει σε μια απόσταση στο Λονδίνο από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στις ε, πολιτικές αυτές άμενας ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής ε, και ασφάλειας. Μεταξύ αυτών των δύο διαφορετικών σχολών και απόψεων πρέπει να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό όμως να καταλάβουμε το λόγο ύπαρξης πίσω από τις δύο τελείως διαφορετικές αυτές σχολές που αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά δύο υπαρξιακές θεωρήσεις εντελώς διαφορετικές σε σχέση με το ποια θα πρέπει να είναι η πεμπτουσία, η βάση της ε, ΚΕΠΑ και της ΚΕΠΑ και τι ε, θέση θα πρέπει να έχει στο ε, όλο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είναι διακυβερνητική η συνεργασία για ενίσχυση ε, των αμυντικών πολιτικών των κρατών μελών, για να είναι πιο αποτελεσματικές, πιο αποδοτικές ε, και για να εξασφαλιστεί περισσότερη ασφάλεια και προστασία για τους πολίτες, ε, αν αυτό θεωρούμε ότι είναι ο ρόλος της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και τίποτε παραπάνω, τότε είναι σαφές. Σε αυτό το πλαίσιο το Λονδίνο πρέπει να παραμείνει στο δυνατόν πιο στενά συνδεδεμένο στην ΚΕΠΑ και την ΚΕΠΑ παρότι ετοιμάστε να αποχωρήσετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, αν θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο αυτό, ότι δεν είναι μόνο ένας διεθνής οργανισμός όπως οι υπόλοιποι, αλλά κάτι παραπάνω, επαναστατικό, ρηξικέλου θα το χαρακτήριζε, το ευρωπαϊκό οικοδόμα είναι επαναστατικό, μια ήρεμη επανάσταση αν θέλετε. Αν θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οργάνωση σου γένερης, υπερεθνική, που έχει μακροπρόθεσμους, βασικούς στόχους, που ε, ένας βασικός στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Όλοκληρία, διακόπτει πάλι η Πρόεδρος. Αν θεωρούμε ότι συνεπεί όλων αυτών η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα, κοινή πολιτική εξωτερική, ε, κοινή εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλεια ε, ακολουθούν την πολιτική που ορίστηκε πριν από 60 χρόνια ε, από τους ιδρυτικούς πατέρες, εάν είναι ένα σχετικό σχέδιο ολοκλήρωσης και όχι απλής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η διασύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου στη λήψη αποφάσεων σε θέματα άμυνας είναι κάτι προβληματικό. Είναι πολύπλοκη, δυσεπίλητη εξίσωση. Πρέπει λοιπόν να κάνει μια επιλογή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχοντας υπόψη την υπαρξιακή θεώρηση που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την αμυντική πολιτική. Το Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο στην πλειοψηφία του υποστηρίζει την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολιτικό σχέδιο ολοκλήρωση και ότι η αμυντική πολιτική είναι μια φάση, ένα στάδιο σε αυτή την χρονοβόρα μακρά διαδικασία ολοκλήρωση, τότε θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Να γίνει σεβαστή δηλαδή εθνική κυριαρχία στου διακανονισμού που θα συμφωνηθούν με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην προκειμένη περίπτωση, η θέση Κομισιόν και Συμβουλίου, κατά την άποψή μου, πρέπει να υποστηριχθεί, να ληφθεί υπόψη. Αν όμω το Κοινοβούλιο αντιλαμβάνεται την αμυντική πολιτική τη Ένωση ω διακυβερνητική συνεργασία για βελτίωση τη ασφάλεια τη Υπήρου και μόνο αυτό, αν δεν έχει δηλαδή κάποιον άλλο από τα το στόχο αυτή η πολιτική, δεν υπάρχει λόγος πράγματι οι Βρετανοί να αποκλειστούν από τη συνεργασία αυτή και για να υπάρχει αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα πρέπει να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν. Η ε, θέση λοιπόν της Κομισιόν είναι ίσως άκαμπτη ε, με αυτή την οπτική γωνία. Στο σχέδιο της μελέτης ε, για το δημοψήφισμα, ακόμη και πιο ε, σκληροπυρηνικοί του Brexit δεν θεωρούσαν ότι θα βγει από το Φόρουμ Ασφάλειας που είναι διακυβερνητικό. Παρόλα αυτά, και δεν ε, έχει μία θέση ευνοϊκή για την ολοκλήρωση, γιατί δεν ήταν ποτέ Βρετανοί Βρετανή και τόσο θετικά διακείμενη απέναντι σε κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον στον τομέα της άμυνας. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η Ένωση είναι ένα σχέδιο ολοκλήρωσης και το λέω ε, για λόγους διαφάνειας, για να μην πει ότι... Ε, δεν είναι κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα μακροχρόνιο σχέδιο ε, ολοκλήρωσης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να είναι πλησωμένη και περιορισμένη η διασύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχωρησή του. Δεν έχω χάσει την ελπίδα μου ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα μπορεί να βασίζεται στο μέλλον περισσότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι αποφασιστική, δεν θα πρέπει να κλείσει παρόλα αυτά και τελείω την πόρτα στο Λονδίνο, που μπορεί να επανέλθει μια μέρα, ίσω όχι αύριο. Κάποια μέρα όμω πρέπει να επανέλθει. Και αν επανέλθει, αυτή τη φορά θα είναι πιο επικοδομητικό, μπορούμε να υποθέσουμε, από τώρα στα θέματα άμυνας. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ακόμη και αν αυτό μπορεί να είναι αφελές. Το Brexit ε, ήταν ίσως αναγκαιότητα στον τομέα της ε, κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και στη ΣΚΕΠΑ και ε, ήταν κάτι απαραίτητο για να ξεμπλοκαριστεί και να προχωρήσει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Οι Βρετανοί όμως ίσως επανειδιοποιηθούν επανικιοποιηθούν στο μέλλον το σχέδιο αυτό και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και επανέλθουν. Οπότε ακόμα πιο πολύ θα αποδειχθεί ότι ήταν αναγκαιότητα το Brexit γιατί ε, ξεκαθάρισε τα πράγματα ε, και έδωσε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, βρει το βηματισμό της. Ποια είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν θέλει να είναι αποφασιστική, ε, πρέπει να είναι αποφασιστική μάλλον, αλλά ταυτόχρονα να μην κλείσει την πόρτα. Πρέπει να είναι το ένα στάδιο να ε, προηγηθεί του δεύτερου. Πρώτα αποφασιστικότητα, μετά ε, άνοιγμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε σε ποιο βαθμό καταρχά το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συνδεθεί στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και σε ποιο βαθμό για να το κατανοήσουμε αυτό νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει ένα σε δύο βασικές ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τη στρατηγική αυτονομία που είναι βασικό, η βασική ιδέα ε, που διαπνέει ότι κάνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διακόπτεται πάλι ο μιλητή. Okay. Σας το έχω πει πολλές φορές μέχρι τώρα ότι μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά συνεχίζετε. Λυπούμε, λέει ο μιλητή. Η στρατηγική αυτονομία είναι ένα θέμα που πρέπει να το απαντήσει η Ένωση για να καταλάβει σε ποιο βαθμό θα πρέπει να συμμετέχουν οι Βρετανοί. Ιδίω τα βιομηχανικά ζητήματα, Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα και μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Αυτά είναι έχω στο μυαλό μου. Η στρατική αυτονομία μπορεί να είναι μέρο τη το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να τεθούν λοιπόν διάφορα ερωτήματα. Μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να θεωρηθεί ένα παράγων που θα πρέπει και θα συνεχίσει να συμβάλλει στη στρατική αυτονομία της Ένωσης. Ναι ή όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, με άλλα λόγια. Πρέπει να είναι από στρατηγική πλευρά αυτόνομη. Με ή χωρί το Ηνωμένο Βασίλειο. Να είναι δηλαδή αυτόνομη και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί σε ποιο βαθμό ε, και μέχρι ποιο σημείο πρέπει να συμμετέχουν οι Βρετανοί στις αποφάσεις ε, για τη μόνιμη διαρθρωμή συνεργασία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Στο Συμβούλιο των Μελών θα πρέπει να συμμετέχουν. Τελικά όμως κάποια στιγμή ε, θα πρέπει να ενταχθούν οι Βρετανοί στις στρατικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με το Ταμείο αυτό. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε λοιπόν στο μέτωπο της στρατηγικής αυτονομίας. Άλλο ερώτημα πώς θα τοποθετηθούν στην Ευρώπη εν γέννη και στον κόσμο οι Βρετανοί. Οι το έχουμε καταλάβει, αρχίζουν σιγά σιγά να ε, είναι κάπως συγκεχημένοι στην απόψή τους για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Έχουν καταλάβει ότι ίσως δεν θα ήταν κάτι αντίθετο με τα δικά τους οικονομικά και βιομηχανικά συμφέροντα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας που προβλέπει τον δεχόμενο κοινωτική προτίμηση που συζήτησε αλλά χρηματοδότηση αμυντικής βιομηχανίας είναι κάτι που ε, προωθείται για να περιοριστούν οι αγορές και εξάρτησή μας από τον αμερικανικό εξοπλισμό. Δεν έχει ε, συμφέρον ε, λοιπόν για βιομηχανική αυτονομία της Ένωσης η Αμερική. Οι Βρετανοί πού θα τοποθετηθούν πάνω σε αυτό. Θα υποστηρίξουν την αρχή της στρατηγικής αυτονομίας στο βιομηχανικό τομέα. Για τους Ευρωπαίους ναι ή όχι πριν καταλάβουμε σε ποιο βαθμό θα του εντάξουμε στην ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να ξέρουμε πώ τοποθετούνται στο θέμα αυτό και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και δεν θα το καταλάβουμε από τη μια μέρα στην άλλη, θα χρειαστεί χρόνο πριν κατανοήσουμε τη θέση των Βρετανών. Προ το παρόν ε, φαίνεται να έχουν πολλά αιτήματα για την ε, πολιτική άμυνας και τη, βιομηχανική, την αμυντική βιομηχανία ε, και εγκομιάζουν σε διάφορα έγγραφα, αλλά το θέμα είναι ε, αν θα παραμείνει έτσι η κατάσταση ε, και αν θα συνεχίσουν να θέλουν την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Σύντομα πρέπει να υιοθετηθεί μια συνθήκη σε θέματα πολιτική άμυνα και βέβαια και για τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα, για να καθισχαστούν οικονομικοί παράγοντε. Είναι σαφέ αυτό. Δεν πρέπει όμω να είναι άκαμπτη η συνθήκη που θα υπογράφει στον τομέα τη Άμυνα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να παραμείνουμε ευέλικτοι. Δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε παραχωρήσει ή να μην κάνουμε. Ανάλογα με τη θέση που θα θετήσει το Ηνωμένο Βασίλειο απέναντι στι διεθνεί αρχέ που μα ενδιαφέρουν. Και θα μετρήσει και η θέση που θα πάρει η Βρετανία όταν κατά πάσα πιθανότητα είπα αρχίζουν λίγο να επαναχωρούν στα θέματα της στρατηγικής αυτονομίας και πολιτικής αμυντικής ε, ε, ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης. Κάτι που ε, αντιστρατεύεται τα δικά του συμφέροντα των Αμερικανών. Επομένως δεν θα πρέπει άμεσα να εγκριθεί μια καμπτή ανελαστική συνθήκη. Χρειάζεται ένα μόνο συνεννόηση, ή ευέλικτες μορφές συμφωνιών. Γιατί έτσι μπορούμε να επηρεάσουμε ε, τη δόση, τη δοσολογία ε, της συμμετοχής ε, των Βρετανών. Και σιγά σιγά να προσπαθήσουμε και να τους επαναπροσεγγίσουμε κοντά στην Ένωση. Ο ιδανικός στόχος θα ήταν να επανέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά με υπευθυνότητα. Ίσως η υπογραφή το συντομότερο δυνατό μια συνθήκη, μια σύμβαση ε, σύνδεση, όπω έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη ασφάλεια και τη άμυνα, ίσω να μην είναι και πλέον ενδεδειγμένη ιδέα. Κατά την άποψή μου, το καλύτερο είναι να παραμείνουν η Ένωση ευέλικτη, να εγκρίνει διάφορε συμφωνίε ε, για του τομεί που σχετίζονται με τον τομέα τη άμυνα ή μνημόνια συνεννόηση και να μην ε, τα βάλει όλα σε άσπρο μαύρο. Ε, και αυτή είναι η πιο βολική λύση γιατί οι Βρετανοί έχουν πολλές απαιτήσει ε, και πολλά αιτήματα. Μπορούμε να κάνουμε ε, υποχωρήσεις και παραχωρήσεις σε κάποια αιτήματα, όλα έχει πάνω στη συμπεριφορά τους. Ποτέ η Ένωση δεν ήταν, αν θέλετε, και τόσο καλά, σε τόσο καλή βολική θέση απέναντι στους Βρετανούς. Γιατί να αλλάξουμε λοιπόν αυτήν την ε, θέση μας. Ευχαριστώ και στο συγγνώμη που μίλαγα τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, ε, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση για τη συζήτηση. Νομίζω να ακούσουμε τρεις-τέσσερις ε, ομιλητές. Παρακαλώ να περιοριστείτε στα δύο λεπτά σε κάθε παρέμβαση και μετά θα ζητήσω από τον κύριο Σαντεπιέτρου να μείνει εδώ στο βήμα και θα καλέσω και τους δύο εμπειρογνώμονες της Κλίνγκελντέιλ, το κέντρο της Ευρωπαϊκής Μεταρρύθμισης που εδρεύει στο Λονδίνο, για να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους για το Brexit και μετά θα γίνει ε, μια πιο μακρά συζήτηση. Αν συμφωνείτε, θα ήθελα να γίνει έτσι η συζήτηση. Καταρχάς ο κύριος Γκάλερ, ο οποίος μάλλον δεν θέλει. Να, θα μπορούσα να αφήσω το λόγο για τον συνάδελφο Ντανζάν. Κύριε Ντανζάν, ευχαριστώ, ευχαριστώ Μιχάλη. με προβλημάτισε λίγο η παρουσίαση που κάνατε αυτή της μελέτη. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, κάποιες απόψεις οι οποίες ε, ομοιάζουν με τις δικές μου, αλλά είναι διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση σε αυτή την προσέγγιση που μας παρουσιάσετε. Θα είχα προτιμήσει να παραμένουμε στα στοιχεία και τους μηχανισμούς που υπάρχουν και πώς μπορούν να λειτουργήσουν αυτοί οι μηχανισμοί χωρίς τους Βρετανούς και πώς μπορούν να λειτουργήσουν και με τους Βρετανούς. Και να σας πω ότι αυτό που με ενόχλησε είναι ότι από τη μια παρουσιάζεται μία διακυβερνητική και μία ολοκληρωτική ε, εκδοχή. Και στα θέματα της άμυνας θεωρώ ότι είναι παράτολμο διότι ποια είναι η θέση της Γαλλίας αυτή τη στιγμή, είναι διακυβερνητική ή της ολοκλήρωσης. Εγώ δεν έχω ιδέα. Υπάρχει η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και των Βρετανών από την άλλη. Και όλα αυτά έχουν διάφορες αποχρώσεις, είναι πολύ σύνθετα και αυτό το οποίο συγκρατώ εγώ είναι ότι σε ένα σύνολο το οποίο όπως πολύ σωστά είπατε είναι σου η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένα οικοδόμημα το οποίο προχωρά με λίγο διακυβερνητικό, με λίγο ολοκλήρωση, με λίγο ε, ευρωπαϊκό και όλα αυτά ε, είναι εύπλαστα ε, η άμυνα είναι ακόμα πιο αεύπλαστο τομέα εντό τη όλη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Να τα κατηγοριοποιήσουμε λοιπόν όλα αυτά έτσι, λέγοντα ότι αν είστε υπέρ τη ολοκλήρωση θα κάνουμε αυτά με του Βρετανού και αν είστε υπέρ του διακυβερνητικού θα κάνουμε αυτά, είναι σαν να περιορίζει τη συζήτηση και τα περιορίζει σε ένα ε, ιδεολογικό ε, πλέγμα το οποίο δεν ε, αρμόζει στη συζήτηση. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ακριβώ το αντίθετο. Θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με του Βρετανού, μπορεί να υπάρχει ένα μόνο κείμενο για την ασφάλεια και την άμυνα, γιατί τα κείμενα που έχουμε για την ασφάλεια και την άμυνα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ελαστικά, πάρα πολύ ελαστικά. Και φανταστείτε τι, πώς θα λέγεται συνθήκη. Ουσιαστικά θα καθορίσει τα πράγματα και νομίζω ότι είναι μια αφηρημένη έννοια. Διότι στα πλαίσια τη ε, πολιτική ασφάλεια και άμυνα. και νομίζω ότι αυτό το λένε και τα κείμενα, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πολύ ευέλικτοι και να είναι τα πάντα πολύ εύπλαστα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα διατηρήσουμε με κάθε κόστο στη σχέση που θα έχουμε με τους Βρετανούς την επαύριο. Και οι Βρετανοί φίλοι μα αυτό το οποίο προβλέπουν για το μέλλον, θέλουν να θεωρούνται ω μια τρίτη χώρα σαν όλου του υπόλοιπου, Δηλαδή μια τρίτη χώρα, σε κάποιες υποψήφιες χώρες ή σε κάποιες ε, χώρες ε, περιθωριακές, περιφερειακές στο οικοδόμημα της ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και νομίζω ότι το να είναι κάποιο τρίτη χώρα στην πολιτική ασφάλεια και άμυνας επιτρέπει πολλά πράγματα. Νομίζω από αυτού συμφωνούμε και στον τομέα της ασφάλειας. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι τρίτη χώρα για κάποιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και κανείς δεν παραβλέπει και τι αντίβαρο έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει πολύ ρεαλισμός, πολύ ευελιξία και θεωρώ ότι είναι ένα κείμενο το οποίο θα εγκριθεί πολύ πιο εύκολα από τα υπόλοιπα γιατί κατά την άποψή μου δεν αποτελεί πρόβλημα θα καθορίσει κάποιες θέσεις και θα αποκλείσει και τριγμούς στο μέλλον. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα σε ένα κείμενο να έχουμε πάρα πολλές ιδέες οι οποίες θα είναι πολύ ελαστικές για το μέλλον και θα επιτρέψουν να έχουν μια σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι προς το συμφέρον όλων. Ευχαριστώ. Η κυρία Κλερμούντι. Ευχαριστώ. Νομίζω μπορώ να πάρω τη σκητάλη από του συναδέλφου Νταντζάν και να συμφωνήσω και θα είμαι και σύντομη, διότι προσβλέπω και στο υπόλοιπο σκέλος της συζήτησης. Συμφωνώ απολύτως ε, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη αναγνωρίζοντας την παρούσα σχέση που έχουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί η μακροπρόθεσμη σχέση, αλλά νομίζω ότι αυτό που με ανησύχησε είναι το τελευταίο σχόλιο σας ε, είναι σαν να λέτε ότι ας περιμένουμε να δούμε, ότι θα πρέπει να το καταπιούμε και αυτό και να περιμένουμε. Ε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Θεωρώ ότι αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο ένα τέτοιο επίπεδο αβεβαιότητας για το πώς θα διαμορφωθεί η συζήτηση δεν βοηθά σε καμία περίπτωση. Ε, να συμφωνήσω δε και με αυτό το οποίο είπε ο κ. Ντανζάν για την ευελιξία που υπάρχει και πρέπει να παραμείνει στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανόρντεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τον ε, καλό συνάδελφο Αρνό Ντανζάν. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε τη μελέτη ακόμα, αλλά εάν το περιεχόμενο της μελέτης αντανακλά τις παρατηρήσεις που μας κάνατε, τότε σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για αντικειμενική μελέτη. Το έγγραφο αυτό θα μπορούσε να βγει απευθεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα κείμενο το οποίο έχει προκαταλήψεις και υποστηρίζει και τις απόψεις ε, τις οποίες ε, ε, πάντα ε, υποστήριζα και εγώ ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα και η ασφάλεια και η άμυνα έρχονται σε δεύτερο επίπεδο. Και φυσικά αυτοί που είναι υπέρ ε, της Ομοσπονδίας, οι φεντερολιστές, είναι πανευτυχείς που αποχωρεί η Βρετανία από το σχέδιο γιατί αυτό θέλανε. Πολλές χώρες στην Ευρώπη πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ προσεκτικά την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Πέραν των στρατιωτικών δυνατοτήτων, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο έθετε περιορισμούς ε, για την ε, δημιουργία αυτόνομων δομών πέραν του ΝΑΤΟ. Δεν αναφέρεται το ΝΑΤΟ καθόλου. Δεν ξέρω αν αναφέρεται ε, στη μελέτη, αλλά η ασφάλεια της Ευρώπης επαφείται στο ΝΑΤΟ και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να συνεχίσει να δεσμεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτού. Επομένως, λοιπόν, και για την Ευρωπαϊκή Έπειρο και για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι προς το συμφέρον όλων να παραμείνουμε στο ΝΑΤΟ. Και ε, η ανησυχία μου είναι ότι επιτρέψαμε να φτάσουν τα πράγματα τόσο μακριά, ιδιαίτερα σε θέματα ανάπτυξη τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Καταρχά, τα 22 κράτη-μέλη της Ένωσης που είναι και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ θα απομακρυνθούν τελικά από την αναζωογόνηση της ε, συμμαχίας που κανονικά θα έπρεπε να είναι προς το συμφέρον όλων και η δεύτερη ανησυχία μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει ακόμα πιο προστατευτική και θα εθελοτυφλή και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ε, συγκεκριμένους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές αναφερθήκατε στον όρο στρατηγική αυτονομία. Ακόμα δεν έχω ακούσει ορισμό για τον όρο, μπορώ να σας δώσω βέβαια τον προσωπικό μου ορισμό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βοηθήσει. Θα ήθελα να ακούσω το δικό σας τον ορισμό. Για να είμαι ειλικρινής όμως δεν νομίζω ότι ήταν αντικειμενική η παρουσίασή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Ερνοντάνζο και την εκτίμηση που έκανε για τη μελέτη σας. Ε, μια πολύ σύντομη διακοπή παρακαλώ συνάδελφοι, ένα λεπτάκι για να έρθουν στο βήμα οι καλεσμένοι μας από το Ινστιτούτο Κλίνγκεντέιλ και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεταρρυθμίσεων και θα συνεχίσουμε με τις δικές τους παρουσιάσεις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 Okay, we are Είμαστε έτοιμοι, οπότε περνάμε στο επόμενο σημείο, αγαπητοί συνάδελφοι, που είναι νομιότυπο με το προηγούμενο, με τη μελέτη δηλαδή που ακούσαμε προηγουμένως, γιατί αφορά και πάλι την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας μετά το Brexit. Με μεγάλη χαρά ε, καλωσορίζω τους επιφανείς μας ε, καλεσμένους, την κυρία Μάργκριτ Ντρέντ, που είναι συντονίστρια της Μονάδας Ασφάλειας στο Ινστιτούτο Κλίνγκεντέιλ, το πασίγνωστο Ολλανδικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Και καλωσορίζω επίσης ε, τον κύριο Ιαν Μποντ, που είναι Διευθυντής Εξωτερικής Πολιτικής στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Μεταρρύθμισης που έχει την έδρα του στο Λονδίνο. Δυστυχώς ο χρόνος είναι ελάχιστος, οπότε χωρίς άλλη καθυστέρηση, κυρία Ντρέντ, ε, σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερος ε, που μπορώ να σας μιλήσω. Το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης ε, εξετάζεται με δύο τρόπους στις ομάδες προβληματισμού και θέλουμε αυτή την διτή προσέγγιση. Καταρχήν το Brexit είναι καλυμμένη ευκαιρία, ευλογία ή καταστροφικό. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί. Σίγουρα είναι προβληματικό το Brexit ε, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει πολλά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια ε, δυνάμεις ε, μεγάλου φάσματος, υπηρεσίες μυστικές με τεράστιες ικανότητες, ειδικές δυνάμεις, αλλά και επιχειρησιακό αρχηγείο. Επίση προσφέρει το 25% των συνολικών οικοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε από άποψη στρατηγικής αυτονομίας, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική αποτελεσματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει αρκετά από, τη, από, το, από το Brexit ε, και θα πληγεί η στρατηγική της αυτονομία. Απ' την άλλη είναι και ένα είδο ευλογία στο Brexit, γιατί όπω ξέρουμε το Ηνωμένο Βασίλειο και η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα δεν ήταν και καλύτερη φίλη μέχρι στιγμής και η δυνατότητα του βέτο που καραδοκούσε σε πολλές πρωτοβουλίες θα εξαφανιστεί πια για το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, το επιχειρησιακό αρχηγείο, η κοινή χρηματοδότηση, η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, η, ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ε, είναι πιο ε, πραγματοποιήσιμα από ποτέ. Και πολλέ άλλε χώρε, ε, όπω και η δικιά μου πατρίδα, η Ολλανδία, πολλέ φορέ κρύβονταν πίσω από την ικανότητα βέτου του Ηνωμένου Βασιλείου, που τώρα θα εξαλειφθεί. Οπότε γι' αυτό έχουμε τη νέα όθηση που έχει δοθεί ε, για την άνθηση της κοινή πολιτικής ασφαλείας και και θα δούμε αν θα συνεχιστεί και αν θα λάβει σάρκα και ωστά. Ε, καταρχήν να αναλύσουμε την συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου στις αποστολές ε, της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που δεν είναι και πολύ εντυπωσιακή δεδομένη ε, της ικανότητας των στρατιωτικών δυνάμεων και του μεγέθους του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάντως, το Ηνωμένο Βασιλείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πολλά κοινά στρατηγικά και αμυντικά συμφέροντα. Και η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια γενικώ έχει πολλά να κερδίσει από μια στενή συνεργασία και στενή σχέση που θα μπορούσε να παραμείνει αλόβητη και μετά τον Brexit. Το θέμα είναι όμως τι μορφή μπορεί να λάβει αυτή η νέα σχέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τρεις κόκκινες γραμμές το Νοέμβριο του 2017. Δηλαδή καμία εξαίρεση για το Brexit, καμία διάκριση εις βάρος τρίτων χωρών δεν έχει λόγο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και επίση αναλογικά δικαιώματα ανάλογα με αυτά που θα προσφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ είναι οι κατευθυντήρε γραμμέ, οι κόκκινε γραμμέ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σημείο φετηρία μα. Εγώ θα έλεγα επίση ότι αυτό που θα προσφέρουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει τουλάχιστον γενικά να μπορούμε να το προσφέρουμε και σε άλλες τρίτες χώρε. Ε, για παράδειγμα, σε ό,τι φορά τη συνεισφορά της Νορβηγίας, δεν θα θέλαμε διάκριση εις βάρος της Νορβηγίας και της ανάμειξης της Νορβηγίας στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Οπότε θα ήθελα στην παρουσίασή μου να επικεντρωθώ σε επιχειρήσεις της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, στην συνεχιζόμενη ανάμειξη σε αυτές, στην χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και στο ΠΕΣΚΟ, τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Αυτή τη στιγμή ήδη ισχύουν πολλές ρυθμίσεις και πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για την ε, βελτίωση αυτών των ρυθμίσεων. Ε, ήδη προσφέρεται μια συμφωνία συμμετοχής και θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον και για τρίτες χώρες. Να είναι ακόμη πιο σε μια τέτοια συμφωνία συμμετοχής για τρίτες χώρες. Επίσης, σε που έχουμε Βρετανούς Αξιωματούχος ε, δεν θεωρείται αρκετή αυτή η συμφωνία. Και το ειδικό καθεστώς που θα επιθυμούσε το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αντικατοπτρίζεται στις ε, παρούσες ε, ρυθμίσεις και διευθετήσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις όντως προσφέρουν από το παρόντος λίγα προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, τα επιχειρησιακά σχέδια, σε διασκέψεις για τη δημιουργία δυνάμεων, απλώς κατόπιν εορτής είναι η συμμετοχή. Οπότε θα διαρωτηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο ή ε, και άλλες χώρες είναι κατάλληλη αυτή η συμμετοχή τρίτων χωρών. Μήπως θα έπρεπε να είμαστε πιο ελαστικοί και μήπως θα πρέπει επ' ευκαιρία του Brexit να εξετάσουμε πιο κριτικά τι προσφέρουμε στις τρίτε χώρε και να αναθεωρήσουμε ίσως και τον τρόπο σκέψη μα ως προς τις τρίτε χώρε. Και σίγουρα δεν είναι σωστό ο παραλληλισμός με το ΝΑΤΟ, αλλά στο ΝΑΤΟ έχουμε πολύ πιο διαφοροποιημένε και βαθύτερες εταιρικέ σχέσεις με τρίτες χώρε. Έχουμε ε, ετε, εταίρους ενισχυμένε εταιρικέ που συμμετέχουν ε, σε διάφορες επιχειρήσεις ε, με ιδιαίτερο τρόπο, αλλά δεν συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και παρόλο που η αυτονομία της λήψης αποφάσεων θα πρέπει να διαφυλαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ θα προτιμούσα μια πιο ε, βαθμία συνεργασία με τρίτες χώρες που έχουν ε, πολιτική και στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, μια πιο σημαντική προσφορά ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας πιο έγκαιρη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ή συνδεδεμένο, καθεστώς συνδεδεμένου μέλους ή καθεστώς παρατηρητή, ανάλογα με το τι συμμετοχή θέλει η χώρα ή το χώρα. Και θα πρέπει να είναι ανάλογο με τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Μόνο έτσι έχει νόημα από άποψη στρατιωτικής αποτελεσματικότητας. Και σίγουρα η κόκκινη γραμμή είναι όχι διακρίσεις και όχι εξαιρέσεις υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, ανταλλαγή πληροφοριών, πολύ σημαντικό στοιχείο της συνεργασίας. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μια συμφωνία για την ασφάλεια των πληροφοριών. Και εδώ όμως ερχόμαστε να με τη δυσκολία ότι η διαιτησία και η άσκηση προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια είναι προαπαιτούμενο που θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε συμφωνία για ε, ρυθμίσεις σε θέματα ασφαλείας. Το ίδιο ισχύει και για τον οργανισμό άμυνας. Από την αρχή ε, ήταν το, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά της αύξησης του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ε, και δεν ε, συμμετείχε πρόθυμα σε σχέδια. Ίσως θα μπορούσε να είναι παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα στη διαμόρφωση της, των αποφάσεων, όχι στη λήψη των αποφάσεων. Το ίδιο ισχύει ε, και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Υπάρχει δυνατότητα συνδεδεμένου μέλους στα προγράμματα πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για τις τρίτες χώρες. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει την αποδοχή της διάταξης για την ελευθερία κίνησης. Ε, ελευθερία διακίνησης και αυτό ίσως είναι πρόσκομα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε πολλά θα πρέπει να εξεταστούν. Και σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης ε, της Άμυνας, και εδώ θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση και αν κάποια μεγάλα επίβολα προγράμματα που απαιτούν την ε, συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου ίσως γίνουν εκτός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην Άμυνα. Αλλά και εδώ προσκρούμε στο θέμα των συμφωνιών που θα έχουμε σε θέματα οικονομικά ή τελωνιακή ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και όσο αφορά τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, την ΠΕΣΚΟ, αυτή θα μπορούσε καταρχήν να είναι ανοιχτή σε τρίτε χώρε για τη συμμετοχή του σε σχέδια. Και επίση πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι αρκετό τρόπο για τη συμμετοχή των τρίτων χωρών στην μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, γιατί οι τρίτε χώρε δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, δεν αποφασίζουν τη στρατηγική κατεύθυνση τη ΠΕΣΚΟ, γιατί αυτή είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά ίσω υπάρχουν ενδιαφέροντα προγράμματα ικανοτήτων ε, στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία και εκεί θα μπορούσαν να γίνουν κάποιε διευθετήσει και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και μέσω του ΝΑΤΟ το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετέχει στα σχέδια στρατιωτική κινητικότητα, για παράδειγμα, στα οποία συμμετέχει, είναι συνδεδεμένο το ΝΑΤΟ. Εν κατακλείδη τώρα κάποιε παρατηρήσεις. Α είμαστε ρεαλιστέ. Αν το Ηνωμένο δεν ενδιαφερθεί να συμμετέχει ε, σε σχέδια ικανοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνα ή τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία ή σε προγράμματα της κοινή πολιτική ασφάλειας και Άμυνα και σε επιχειρήσεις και αποστολέ, τότε θα λάβει πολύ λιγότερα προνόμια και δεν θα έχει τόσο λόγο στην διαμόρφωση των αποφάσεων ενδεχομένω. Οπότε ελαστικές ρυθμίσεις, μια προοδεστική βαθμία συνεργασία θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο για, για τις τρίτες χώρες και αν το Ηνωμένο Βασίλειο ενδιαφέρεται για συνεργασία και ενίσχυση της συνεργασίας στο CSDP, στην κοινή ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας, τότε μια τέτοια βαθμία σχέση θα είχε νόημα και ουσία. Ευχαριστώ. Αυτά. Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ιαν Μποντ, το Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεταρρύθμισης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι σήμερα το πρωί εδώ. Η πρώτη, ίσως και η τελευταία φορά είναι αυτή που μου δίνεται η δυνατότητα με την επικείμενη αποχώρηση. Αυτό που θα ήθελα να κάνω σήμερα είναι να πω λίγα λόγια <clears throat> για το σημερινό ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στην ε, ΚΕΠΑ και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Για να δούμε τι σχέσεις θα ήθελε ενδεχομένω η Βρετανική κυβέρνηση μετά το Brexit. <clears throat> Μετά θα σας αναφέρω τις ανησυχίες μου για την πολιτική ασφάλεια και άμυνας που θα ήθελε η Ένωση να ακολουθήσει μετά το Brexit και τέλος θα καταλήξω με κάποιες συστάσεις για το πώς θα αποφύγουμε να βλάψει σημαντικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα το Brexit. Καταρχά, επειδή το είπαν προλαλήσαντε ομιλητέ, πρέπει να αναγνωρίσω ότι κατά το παρελθόν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ένα εμπόδιο στην αμυντική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχώς προτιμούσε το πλαίσιο ε, του ΝΑΤΟ η δημερή συνεργασία με συμμαχίες προθήμων, τη ΣΥΠΑ, έχει μπλοκάρει διάφορες πρωτοβουλίες όπως το επιχειρησιακό στρατηγείο, κατάφερε τον προπολισμό του Οργανισμού Άμυνας να τον διατηρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν ήταν καθόλου ενθουσιώδες σε ό,τι αφορά ε, την οδηγία για τις προμήθειες ε, στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών όταν συζητεί το, το θέμα αυτό. Πάντως ε, φάνηκε με τη Συμφωνία του Καλοκαίρι ότι χρειά ε, θα, θα δώσει τη σύμφωνη γνώμη του το Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν υπάρχει βέβαια ε, ανταγωνισμός με τον ΝΑΤΟ, θα παρέχει το επιχειρησιακό στρατηγείο για την Αταλάντη και αν δει κανεί τα στατιστικά, μετά την οδηγία, ε, τη θέση ισχύ τη οδηγία για τι δημοσίε προμήθειε, κανένα κράτο μέλο δεν την αξιοποιεί τόσο όσο το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο, εν γέννη, συμμετέχει ενεργά ε, στην ε, κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Είναι ο τρόπος τρόπο που προτιμά για να επιδιώξει του στόχου του το Ηνωμένο Βασίλειο. Στα τέλη του 1996 είχα και εγώ βοηθήσει να καταρτιστεί το πρώτο σχέδιο της κοινή θέση της Ένωσης για το Αφγανιστάν και την Κούβα. Υπό συντηρητική κυβέρνηση που ήταν προσκεπτικιστική σε άλλες ε, πτυχές. Άρα υπάρχουν πράγματα πιστεύω όπου το Ηνωμένο Βασίλειο παρότι ενίοτε χρησιμοποιεί ρητορική ε, αντιευρωπαϊκή, στην πράξη ήταν ενεργό και χρησιμοποίησε τους ε, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Τι σχέση λοιπόν θέλει για το μέλλον του ΕΒ. Βασίλειο. Η κυβέρνηση δεν έχει μπει σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας, προς το παρόν αλλά είναι σαφές ότι θέλει πιο στενές αμυντικές σχέσεις από οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα με την Ένωση στη διάσκεψη ασφάλειας του Μονάχου το Φεβρουάριο είπε η Τερέζα Μέη ότι είναι ανοιχτό το Λονδίνο να συνεχίσει να συνεισφέρει στις επιχειρήσεις ή ε, αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν σαφής επίσης η κυβέρνηση ως προς το ότι θα ήθελε ε, να συμμετέχει και στον αναλυτικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων και την κατάρτιση των εντολών. Αυτό είναι προϋπόθεση για να δώσει και στρατεύματα. Το Ηνωμένο στη συνέχεια αυτό είναι αμφίδρομο βέβαια. Δηλαδή θέλει να έχει λόγο το Ηνωμένο Βασίλειο για να ε, συνεισφέρει. Η κυβέρνηση θέλει να βρει σίγουρα έναν τρόπο να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και ελπίζει 27 της Ένωσης ε, να έχουν μια ανοιχτή προσέγγιση που να είναι υπέρ της συμμετοχής των Βρετανών στην ανάπτυξη δυνατοτήτων. Ένα άλλο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενδιαφέρεται να καταλήξει σε συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής ε, που θα εφαρμόζεται κατά τη μεταβατική περίοδο μετά το Μάρτιο του 2019, χωρίς να περιμένει την τελική συμφωνία, όποια και αν είναι αυτή, που θα ισχύσει στα τέλη του 2020. Και αυτό νομίζω ότι αντικατοπτρίζει και την ε, δύσκολη θέση, την αμηχανία του ε, Ηνωμένου Βασιλείου να δεσμεύεται από τι αποφάσει Ευρωπαϊκή Ένωση για του πολύ δελπτού και ευαίσθητου τομεί για την εθνική ασφάλεια και εθνική κυριαρχία τομεί. Όταν θα έχει χάσει τη φωνή του ε, στου φορεί λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να πω ότι αυτό που με ανισχύει εμένα περισσότερο είναι η κατεύθυνση στην οποία θα οδηγηθεί ενδεχομένως η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας ε, στην Ένωση μετά το Brexit. Δεν νομίζω ότι θα ε, συρθεί από αδίστακτη μιλταριστική Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολέμους ε, στην Αλλοδαπή, το Ηνωμένο κάτι που ως επιχείρημα χρησιμοποίησαν οι ευρωσκεπτικιστές το 2016 και το συσχέτισαν με την εμπεριληστική πολιτική της Ένωσης στην Ουκρανία, για παράδειγμα. Αυτό που με ανησυχεί λοιπόν πολύ είναι ότι μετά το Brexit, η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως ε, γίνει πιο πολύ παρατηρητής, παθητικός παρατηρητής ε, στα τεκτενόμενα στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας. Ακόμη και με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ανησυχώ. Μήπως η Ένωση δυσκολευτεί να κλείσει τα κενά στις δυνατότητες και να αποκτήσει μια στρατηγική κουλτούρα που οι προκλήσεις σήμερα στην ε, Ευρώπη ε, απαιτούν στον τομέα της ασφάλειας. Επί το παρόντος, με εξαίρεση τη Γαλλία, λίγα, πολύ λίγα είναι τα κράτη-μέλη που παίρνουν σοβαρά, αρκετά σοβαρά ε, υπόψη τους την άμυνα. Δεν μιλάω για τον αμυντικό προπολογισμό του 2% ε, που είναι ένα συμβολικό ποσό. Αλλά δεν είναι και αυτός σκοπός. <clears throat> Το θέμα είναι να έχεις δυνάμεις επιτόπου που μπορούν να αναπτυχθούν, να αντιμετωπίσουν διαφορετικού είδους απειλές σε διαφορετικούς τόπους. Επίσης ε, μιλώ για πολιτικούς που θα έχουν την προθυμία να πάρουν δύσκολες αποφάσεις ε, και να βάλουν σε κίνδυνα στρατεύματα και να ε, αιτιολογήσουν και στους ψηφοφόρους τους γιατί είναι ότι χρειάζεται να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις και επίσης ε, πρέπει να λαμβάνονται και αποφάσεις σε σχέση με τις προμήθειες για την απόκτηση του καλύτερου δυνατού εξοπλισμού στην καλύτερη δυνατή τιμή όχι μόνο στα πανηρό τρόπο υποστήριξης της απασχόλησης στις μονεκτικές περιοχές. Και ξέρω ότι υπάρχουν πιέσεις σε κάποιες χώρε περισσότερες από άλλες, αλλά ε, όταν έχουμε ε, πρόβλημα ε, λιτότητα με τους προπολογισμού, καλό είναι να εξοπλίσουμε το κάθε ευρώ στον τον περισσότερο. Πώς θα περιορίσουμε τις ζημίες λοιπόν από τον Brexit. Προσωπικές μου σκέψεις. Το σημαντικό είναι ότι οι 27 της Ένωσης δεν θα πρέπει να βλέπουν το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο ε, με τα γυαλιά ε, της παλιάς του συμπεριφορά στη διεθνή συνεργασία, θεωρώντας ότι καλύτερα να μην είναι στην Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί έχει σημαντική στρατιωτική συνεισφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι πάντα στις επιχειρήσεις της πολιτική πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, αλλά θυμάμαι ότι όταν ξεκινούσαν, δρομολογούνταν πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις, Ευρωπαϊκή, το Ηνωμένο Βασίλειο έδινε πολλά στρατεύματα, ιδίως για το Αφγανιστάν. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προηγμένο ε, αμυντικό βιομηχανικό τομέα που μπορεί να βελτιώσει την άπτυξη ε, δυνατοτήτων της Ένωσης να του επιτρέπει κάτι τέτοιο. Και ναι μεν μπορεί να είναι πειρασμό να πει κανεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οποιαδήποτε τρίτη χώρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν δεν το θέλει αυτό για τον εαυτό τη ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν καλό να αντισταθούν στον πειρασμό 27. Κατανοώ τις πολιτικές ε, επιπλοκές στο να γίνουν διακρίσεις μεταξύ των διαφορετικών ευρωπαϊκών, νατοικών χωρών και χωρών μελών του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλη της Ένωσης όμως. Κατανοώ τη δυσκολία, αλλά υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ μιας χώρας που είναι ή ήταν μέλον της Ένωσης και συνεισέφερε στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής και εξακολουθεί να θέλει να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Υπάρχει μια διαφορά από αυτή τη χώρα, μεταξύ αυτής της χώρας και των άλλων. Θα πρέπει νομίζω να αναγνωρίσουμε τις δυνατότητες που μπορεί να παράσχει για επιχειρήσεις η ε, Βρετανία. Βρετανική δέσμευση ε, μέσων στρατευμάτων σίγουρα θα απαιτεί διαβούλευση και ανταλλαγή πληροφοριών στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά την αμυντική έρευνα και τις δημόσιες προμήθειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πρόθυμη να επιτρέψει σε βρετανικές οργανώσεις ε, να ε, κάνουν έτοιμα για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεχίσουν τη ρυθμιστική ευθυγράμμιση με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν τι διμερού σχέσει αν θέλετε, μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελπίζω οι χαράκτε πολιτική Ένωση να δώσουν προτεραιότητα και στο μέλλον στι στενέ σχέσει με τον ΝΑΤΟ. Πολύ πρόοδο σημειώθηκε μετά την κοινή διακήρυξη τη Βαρσοβία το καλοκαίρι του 2016. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονό ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει όχι μόνο στρατιωτικέ απειλέ σήμερα, πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό της ε, η Ευρώπη, αλλά κάποιε περιπτώσεις αυτό είναι στα χέρια του ΝΑΤΟ, κάποιες είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 22, 21 χώρες είναι μέλη και των δύο οργανώσεων και η συνεργασία τους ε, είναι κάτι ζωτικής σημασίας. Ολοκληρώνοντας, δύο λόγια για τη στρατιωτική κουλτούρα που θα πρέπει να κρατήσει μετά τον Brexit η Βρετανική κυβέρνηση. Μάλλον οι Βρετανικέ κυβερνήσει και των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων ε, παραδοσιακά δέχονται ότι η χρήση βία δεν είναι ευκταία, αλλά ίσω εννοεί ότι είναι ο μόνο τρόπο να αντιμετωπιστούν κάποιοι παράγοντες που θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους εξωτερική πολιτική με τη χρήση της βίας ε, και αυτό τους είναι πολύ πιο εύκολο από ότι είναι σε εμά. Ίσως είναι άποψη με ψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που θα πω, αλλά κάθε φορά που ακούω την είπατε εκπρόσωπο ή άλλους να λένε για κάποιες συγκρούσεις αντιπαραθέσεις ότι δεν υπάρχει στατιωτική λύση ε, σε αυτήν την αντιπαράθεση ε, προβληματίζομαι εντόνως. Πάντοτε υπάρχει στατιωτική λύση και κάποιοι είναι έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσουν. Μπορεί για ιστορικούς ή άλλους λόγους τα τα κρατη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κάποιες εξαιρέσεις, να χρειαστεί να ακολουθήσουν πια πιο βρετανική ε, προσέγγιση όταν φύγουν οι Βρετανοί. Να γίνουν Βρετανοί στη θέση των Βρετανών. Αν χρειαστεί να υπερασπιστεί αυτόν η Ένωση, θα πρέπει να δείξει ότι είναι έτοιμη να κάνει χρήση βίας αν αυτό καταστεί αναγκαίο. μην είναι δηλώσεις, κυρώσεις ε, που δεν θέλουν όμως να ε, δημιουργήσουν πρόβλημα σε εμάς αλλά στους αντιπάλους δεν αρκούν. Και εδώ σταματώ. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσει η συζήτηση ο κύριος Γκάλερ πρώτα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω με αυτό με το οποίο συμφωνώ, που είναι ένα από τα τελευταία που αναφέρατε. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ευχόμαστε ένα καλύτερο κόσμο από ότι είναι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα ως έχει και να λάβουμε μέτρα τα οποία είναι κατάλληλα δεδομένων των συνθήκων. Και νομίζω ότι στην ίδια με τη χώρα, στη Γερμανία, θα πρέπει να γίνουν σοβαρές συζητήσεις επί του θέματος, προκειμένου να μπορέσουμε να σταθούμε και στο ύψος των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επιπλέον, πρέπει να πω ότι θα ελέγξουμε διεξοδικά τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Και αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι η Βρετανία τώρα που αποχωρεί ε, φαίνεται να αναζητάνε ε, απελπισμένα και ε, μεθόδους συνεργασίας. Βέβαια υπάρχει η φράση ότι κάποιος ε, που αποχωρεί δεν μπορεί να είναι σε καλύτερη κατάσταση ε, ή έστω και στο ίδιο επίπεδο με αυτούς που ε, παραμένει. Έχω μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, την Νορβηγία, και έχω και μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, τη Βρετανία. Η Νορβηγία είναι και στη Σέγγεν και σε άλλες συνθήκες. Και η Νορβηγία αξίζει καλύτερη συμπεριφορά, διότι είναι πιο ενταγμένη. Πέραν αυτού, είμαι διατεθειμένος και να ελέγξω πώς μπορούμε με ρεαλιστικό τρόπο να οργανώσουμε τη μελλοντική συνεργασία. Όταν λέτε ότι έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε, ναι μεν, αλλά ε, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από τις, στις αποστολές ε, ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας στο παρελθόν και σε ποσοτικούς όρους. Δεν ε, το είδαμε αυτό μέχρι τώρα στο μέτρο του δυνατού. Όσον αφορά λοιπόν τους τομείς της βιομηχανικής συνεργασίας, υπάρχει νομοθετική πρόταση EDTP στα σκαριά. Και η προσέγγιση μου ήταν σε έκτακτες περιπτώσεις και αν υπάρχει παραγωγή στη χώρα μας και αν πληρώνετε τους φόρους σας και δεν υπάρχουν και νομικά κολλήματα για τη χρήση των προϊόντων τα οποία διαθέτουμε, τότε ίσως θα μπορούσε να υπάρχει και συμμετοχή αν συμβάλλεται και αυτό το οποίο προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση. Ε, ναι, σαφώς λοιπόν υπάρχουν δυνατότητες στον τομέα αυτό, αλλά δεν μπορούμε να είναι όπως ε, ήταν ε, στην περίπτωση που θα παραμένατε. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχουμε 12 λεπτά το πολύ. Η κυρία Μούντι. Ευχαριστώ. Και πάλι θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Πιστεύω ότι είναι και κρίμα που ο συντάκτης της μελέτης... Α, εδώ είστε, συγγνώμη. Ίσως λοιπόν να είναι χρήσιμη και η συμβολή για την εξέλιξη της συγκεκριμένη μελέτης ε, τα όλα όσα ακούσαμε τώρα. Και νομίζω Αυτά τα οποία θα πρέπει να δούμε μαζί με το Brexit είναι να προσπαθήσουμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες όπως έχουμε τώρα να ε, τα πετάξουμε όλα και να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Αναγνωρίζω βεβαίως ότι υπάρχει ευθύνη του Ηνωμένου Βασιλείου, της κυβέρνησης ε, να κάνει επικοδομητικές προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το μέλλον, αλλά υπάρχουν και πράγματα που όντως μπορεί να συμβάλλει το Ηνωμένο Βασίλειο στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι δεν θα πρέπει όλα αυτά ε, να τα διακόψουμε και να τα πετάξουμε στα σκουπίδια. Ε, θεωρώ ότι είναι ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ε, συμφωνία γέρος αρκετά νωρίς, στο μέτρο βεβαίω του δυνατούν και αυτό κατά την άποψή μου θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και φυσικά το σχέδιο της ασφάλειας και άμυνας που είναι αυτό το οποίο συζητούμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κάρβερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ βέβαια είμαι υπέρμαχος του Brexit, επομένως έχω τελείως διαφορετική προσέγγιση από ό,τι έχουν κάποιοι συνάδελφοι εδώ στην αίθουσα. Η άποψη του κυρίου Γκάλερ ε, μου φαίνεται και λίγο απερπισμένη. Στα τέσσερα χρόνια που είμαι πλέον εδώ στο Κοινοβούλιο, βλέπω ότι προσπαθούσαμε να συζητήσουμε με τον συντονιστή και όταν δέχτηκε να μιλήσει μαζί μας, και αυτά ήταν πολύ πριν τα δημοψηφίσματα και το Brexit, είδαμε πόσο ε, βασίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και για την... Ε, ε, ε, ανταλλαγή πληροφοριών και για πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή ε, πρέπει να τα δούμε αυτά συγκεκριμένα. Αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Άμυνα ή στην Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με όλο το σεβασμό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τα βλέπει υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένας και όχι τα δικά του εγωιστικά συμφέροντα και μόνο. Έχουμε το ΝΑΤΟ φυσικά, ο κύριος Ντανζάν, ο φίλος και ο συνάδελφος από το ΕΛΚ, ε, να θυμάμαι και τις ε, συμφωνίες ε, που έκανε η χώρα μου με τη Γαλλία το 2010. Έχουμε και κοινέ αποστολές, το JEF, με σκανδιναβικές χώρες και χώρες της Βαλτικής. Και από ό,τι βλέπουμε, αυτές λειτουργούν αποτελεσματικά σε διμερές επίπεδο, σε, πολλές, σε πολλά μέτωπα. Και γιατί όχι άλλωστε. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε, και εγώ μιλάω από ε, το πρέσμα κάποιου που ήμουνα υπέρ της Ευρώπης και άλλαξα τη γνώμη τελικά, πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι ευρωπαϊκό. Φαίνεται σαν να μας αρέσουν οι ξένοι, σαν εγώ να έχω ε, πρόβλημα με τους Πολωνούς, ε, για παράδειγμα. Τι γίνεται όμως για την, με την ουδετερότητα, για παράδειγμα, της, και άλλες χώρες, την Αυστρία, τη Σουηδία. Συγγνώμη, πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να είστε σύντομος και ο κύριος Μπόρν έκανε ένα σχόλιο και τελειώσατε με πολύ ε, καλό τρόπο και σας συγχαίρω για αυτά που είπατε. Το Brexit ουσιαστικά, όπως είπε και ο κύριο Γκάλερ, είναι η στιγμή στην οποία τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν τι ευθύνε έχουν. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την ουδετερότητα, την οποία θίξατε ακροθυγώς. Ευχαριστώ κύριε Ντανζά. Έχω κάτι το οποίο θα πω σύντομα, δεν θα επαναλάβω τα προηγούμενα, διότι πιστεύω ότι η περίοδος μετά το Brexit είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε χωρίς δράματα στο θέμα αυτό. Υπάρχει αμοιβαία συνεννόηση ούτως ή άλλως, ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Υπάρχει λοιπόν και ρεαλισμός και ευελιξία για να τα καταφέρουμε στο Brexit. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω και με ένα ψήγμα ηρωνίας κάποιες ε, βρετανικές θέσεις οι οποίες με κάνουν να μη διάζω τη σήμερα ημέρα. Πολλοί Βρετανοί φίλοι μας λένε σήμερα «Α, δεν ξέρετε τι χάνετε σε θέματα άμυνας ε, και ασφάλειας με τον Brexit». Ναι, δεν ξέρουμε, γιατί οι Βρετανοί μέχρι τώρα δεν μας είπαν και πολλά για το τι θα μπορούσαν να συμβάλλουν ε, λένε ότι α, συνεισφέραμε πολύ στην ΚΕΠΑ και όχι την ε, πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Α, ναι, συνεισφέρατε πολύ. Στατιστικά δεν είναι αποδεδειγμένο αυτό και θα σας περιγράψω και μια συζήτηση που είχαμε έναν Υπουργό ε, Άμυνας Βρετανό πριν από λίγο καιρό που μου έλεγε κύριε Ναζάν φαντάζεστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει κάτι φιλόδοξο σε επίπεδο ναυτικού χωρίς το πολεμικό ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου. Ναι φυσικά την αποστολή Αταλάντα. Ε, δεν υπήρχε κανένα βρετανικό σκάφος που να συμμετείχε στις περιπολίες κατά της πειρατείας ε, στις ακτές της Ομαλίας. Και όλοι θεωρούν την επιχείρηση Αταλάντη επιτυχημένη. Έχουμε λοιπόν ένα παράδεξο. Ναι, σε απόλυτε τιμέ, ε, πράγματι το Ηνωμένο Βασίλειο σε επιχειρησιακές δυνατότητες είναι ε, μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη. Αλλά όσον αφορά την πραγματική συμβολή της ε, στην ΚΕΠΑ είναι ισχνά ε, τα όσα έχει κάνει. Πάρα πολύ συχνά και πραγματικά μου φαίνεται ηρωνία να έρχεται κάποιο να μου λέει ότι θα χάσετε, όταν στην πραγματικότητα δεν έχει συμβάλει και πάρα πολλά το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τώρα. Ε, όσον αφορά τις διμερεί συμφωνίες, σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες διμερέ πτυχέ, οι οποίε θα είναι αρκετά έντονε, κυρίω ο αγγλογαλλικό άξονα είναι πολύ σημαντικός. Να πω και στο φίλο Κάρβερ ότι η πιο μεγάλη επιχείρηση στην οποία έχουν δεσμευτεί ευρώ δεν είναι ευρωπαϊκή επιχείρηση, αλλά συμμετέχουν περισσότεροι οι Ευρωπαίοι, είναι στο Σαχέλ. Ε, ε, Γερμανοί, ε, Ολλανδοί, Σουηδοί, σε διάφορες συνθέσεις. Ε, στην ΙΜΣΜΑ, στην, από πλευράς Αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Βρετανοί έχουν συμβάλει τρία συνούκ. Εντάξει, είναι σημαντικό, αλλά μην θεωρείτε ότι είναι εκεί η μεγαλύτερη συμβολή. Είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση στην οποία δεσμεύεται και τι έχουν δώσει τρία ελικόπτερα. Ε, θα ήθελαν να συνεισφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά στην πράξη δεν ισχύουν όλα αυτά. Thank you. Σας ευχαριστώ ο κύριος Γιάννος Ζέμκε, μα δεν μας έμεινε χρόνος, οπότε επιγραμματικά μόνο τηλεγραφικά και μετά θα κλείσω τον κατάλογο των αγορετών. Γιατί πρέπει να δώσουμε το λόγο και στους Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ένα μόνο πράγμα. Αν περιμένουμε, περιμέναμε άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, έχουμε τώρα το φαινόμενο ότι οι πολίτες μας περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει περισσότερες ευθύνες για την ασφάλεια των πολιτών. Αυτό είναι το νέο φαινόμενο. Και η ερώτησή μου είναι η εξή. Στον το με αυτό θα μπορούσαμε, θα περιμένουν οι πολίτες να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ θεωρώ πως ναι. Και θα πρέπει να σκεφτούμε τι είδους συγκεκριμένες συνεργασίες και συγκεκριμένες δράσεις μπορούμε να έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο και από στρατητική άποψη και από άποψη ανταλλαγής πληροφοριών και νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ιδεολογία αλλά έμπρακτες μορφές συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Λυπούμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. 1,5 λεπτό μόνο στον κύριο Σαντοπίντο για να απαντήσει. 1,5 λεπτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, για να απαντήσετε σύντομες παρατηρήσεις που έγιναν προηγουμένως από τους συναδέρφους και κατόπιν πολύ σύντομα επίσης τους ε, άλλους δύο καλεσμένους μας. Δυστυχώς, κυρία Πρόεδρε, οι περισσότεροι ευρωβουλευτές που επέκριναν την ε, μελέτη μου αποχώρησαν στο μεταξύ. Ευχαριστώ όμως τον κύριο Ταζόν που παρέμεινε. Εύστοχη κριτική του. Κύριε Ντανζόν. Είπατε ότι δεν θα πρέπει να ε, έχουμε αντιπαράθεση μεταξύ της αντικυβερνητικής προσέγγισης και της προσέγγισης της ολοκλήρωσης. Ναι, μεν, αλλά αν ε, θέλουμε μια πολιτική άμυνας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος. Και ο λόγος είναι ότι αυτό το πολιτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής ε, Άμυνας θα πρέπει αργά ή γρήγορα, ίσως όχι τώρα αμέσω, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον, θα πρέπει να ταχθεί σε ένα ευρύτερο σχέδιο. Ε, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σχέδιο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δεν λέω ότι θα πρέπει να είναι φεδεραλιστικό κατά ανάγκη. Αλλά το γεγονό ότι η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα γίνεται εντό και όχι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γιατί ε, μακροπρόθεσμα θα ενταχθεί στο ευρύτερο σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, γιατί θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αποδώσουμε μια Ευρωπαϊκή Άμυνα. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να βάλετε τελεία. Και τώρα πολύ σύντομα παρακαλώ η κυρία Τρέντ και μετά ο διευθυντή ο κύριο Μποντ. Λυπάμαι, αλλά δυστυχώ μα πιέζει αφόρητα ο χρόνος. Πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε τέτοιου είδου συζητήσεις και συνεδριάσεις. Ευχαριστώ, όντως είναι πολύ εύλογο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσπίσει τα αμυντικά της, τα συμφέροντά της ασφάλειας γιατί υπάρχει μια επιδείνωση στην ασφάλεια και θα πρέπει να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα ενισχύσει την ασφάλειά της και ήταν επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα πρέπει να βρούμε τρόπο να αναμίξουμε ε, στο μέτρο του δυνατού το Ηνωμένο Βασίλειο στις προσπάθειές μας και θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ε, να δούμε τι περιβάλλον ασφάλεια έχουμε, ποιο είναι το τοπίο τη ασφάλεια και αν θέλουμε να είμαστε σημαντικό παράγοντα στον τομέα τη ασφάλεια, ε, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί υπάρχουν και άλλε συνασπισμοί και άλλε συμμαχίε που χρησιμοποιούνται περισσότερο για να αντιμετωπιστούν οι απειλέ στην ασφάλεια. Πάντω θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε ρεαλιστέ, πραγματιστέ και να αναμίξουμε το Ηνωμένο Βασίλειο όσο περισσότερο γίνεται σε αυτά τα σχέδια. Σα ευχαριστώ. Ο Διευθυντή ο κ. Ιαν Μποντ. Σα ευχαριστώ συμφωνώ πλήρω με τον κύριο Ντανζό για την περιορισμένη συμμετοχή, συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου στις αποστολές ε, ε κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ε, πολλά μπορεί να γίνονται πιο διακριτικά στα παρασκήνια, αλλά μακάρι να ήταν πιο ορατή η συμμετοχή. Και τώρα ε, φαίνεται να ανα, αναφέρεται μεγαλύτερη ανάγκη συμμετοχή τώρα που φεύγουμε. Κύριε Κάρβερ, σίγουρα υπάρχουν πολλοί τρόποι με του οποίους μπορεί να παραμείνει ενεργό σε θέματα ευρωπαϊκής άμυνας το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι κάποια επιθυμητή συνεργασία ε, επιδεινώνεται λόγω της αποχώρησης. Και γι' αυτό και η ε, συμμετοχή και η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμη πιο σημαντικές στο μέλλον, γιατί οι ε, απειλέ είναι όλο και περισσότερες και δεν εμπίπτουν στις παραδοσιακές ε, μέχρι στιγμής δράσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο της σα διάταξης και ευχαριστώ θερμά τους εμπειρογνώμονές μας και να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να μεταβούμε στην αίθουσα 3Ε2 στο κτίριο Αλτιέρο Σπινέλη για το στρατηγικό διάλογο με την Φεντερίκα Μογκερίνη. Και θα επανέλθουμε στην ίδια αίθουσα εδώ στις 11 που θα ακούσουμε τον αντιστράτηγο Λούδη Κλάιν Χάους που είναι επικεφαλής του Κέντρου Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο ε, της Γερμανίας. Ευχαριστώ.